Κυρίε και κύριοι, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη για απόψε. Γρήγορε ανακοινώσει. για τη μετάδοση στο διαδίκτυο. Δεν είναι πολύ καλό το προηγούμενο βέβαια, αλλά λόγω τεχνικών περιορισμών θα ηχογραφηθεί η συνεδρίαση και θα διατεθεί αργότερα διαδικτυακά. Η Γερμανία θα υπάρχει σε όλες τις γλώσσες εκτός των εστονικών, των λιθυνανικών, των κρατικών και των γελικών. Να καλωσορίσω τους συναδέλφους και των δύο επιτροπών της ΙΜΚΟ και της ΙΤΡΕ, οι οποίοι συνεργάστηκαν τόσο αρμονικά για την έκθεση αυτή και ορισμένους αναπληρωτές επίσης να σας θυμίσω ότι ήταν 1287 οι τροπολογίες ε, στην έκθεση, χωρίς να μετράμε τις νομοδοτήσεις των υπολείπων επιτροπών. Θα, θα συγχαρώ θερμά λοιπόν και την κυρία Κάλλα τη Επιτροπή Ήτρε και την ε, κυρία Γκέπχαρτ από την Επιτροπή ΙΜΚΟ και του κοιόδη συζητητέ και των δύο ε, επιτροπών για την απίστευτα σκληρή δουλειά του και την φοβερή του συνεργασία με τόσε πολλέ συναντήσει και συνεδριάσει να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες, μου, συνεργάτες μας από τη Γραμματεία, τους συμβούλους και βοηθούς, οι οποίοι επίσης ε, εργάστηκαν και μέχρι εργά τα βράδια για να φτάσουμε στη σημερινή ψηφοφορία. 54 είναι οι συμβαστικές τροπολογίες και διερωτώ με αν εάν αυτό θα αποτελέσει και το, την πορεία της ψηφοφορίας, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Να συγχαρώ και τους ε, σκέωτες και τους εισηγητές των υπολείπων επιτροπών που έφεξαν πολύ μεγάλο ρόλο, ιδίως στις τελευταίες συναντήσεις των σκεωδών, ώστε να συνδυαστούν όλες οι τροπολογίες. Θα πρέπει να μας πάρει δυόμιση ώρες λογικά περίπου η ψηφοφορία, αλλά ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπετε. Να δώσω το λόγο και στον συμπρόεδρο, τον Γιέρζη Μπούζεκ, με τον οποίο ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Βίκη. Πραγματικά είχαμε συνεργατικούς σχηματισμούς υπέροχους, φανταστικούς, 8 επιτροπών και 6 επίσης πολύ στενές μορφές συνεργασίας σε στενή επαφή με τις δύο καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές. Αυτή είναι η απόκρισή μας για τη νέα μορφή σχηματισμού και εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για την ενιαία ψηφιακή αγορά και για την ε, ψηφιακή ένωση. Στο μέλλον θέλουμε να οικοδομηθεί μια ψηφιακή ένωση. Δύσκολο αλλά πολύ σοβαρό το θέμα, το όλο το σχέ, το ξέρουμε πολύ καλά και η πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και η Δίκη, μεταξύ και των έξι επιτροπών ήταν πολύ ε, αποτελεσματική. Οι δεν ήταν ποτέ εύκολη, όπως ξέρετε, αλλά παρόλο που είναι μακρό, μακριοσκελής ο κατάλογος των ψηφοφοριών, ελπίζω να τα καταφέρουμε πιο γρήγορα από ό,τι θα περιμέναμε. Καλή μας τύχη λοιπόν για την επόμενη ώρα και 20 λεπτά. Δεν είναι αγώνας δρόμου, αλλά θα προεδρέψω στο πρώτο ίμιση της ψηφοφορίας και στο δεύτερο ο κύριος Μπούζεκ. Και έτσι ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια εύρυθμη διαδικασία. Αν μπορούμε γρήγορα να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 1ης Δεκεμβρίου, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και δεν υπάρξουν στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν. Προχωρούμε λοιπόν στην ίδια την ψηφοφορία και να σας θυμίσω ότι έχουμε 180 ψηφοφορίες συνολικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλώς να θυμίσω, όπως μου σημείωσε και η Γραμματεία, ότι η τροπολογία 396 δεν καλύπτεται από την συμβιβαστική 14α. Οπότε θα ψηφιστεί ξεχωριστά. Έχει ειδοποιηθεί η γραμματεία και πρέπει να έχουν διορθώσει αναλόγως και τον κατάλογο. Η γραμματεία μου λέει ότι θεωρεί ότι η τροπολογία σας 396-396 καλύπτεται από, τον, από τη συμβαστική 14α συγχωρείτε. 3B. 3Β για την πολιτική ανταγωνισμού. Η τροπολογία σε 396 αφορά την πολιτική ανταγωνισμού και θεωρούν ότι ουσιαστικά τμήματα της τροπολογίας σας καλύπτονται έτσι και από την συμβαστική 3B. 3B για, την, ε, για τους νόμους του ανταγωνισμού. Άλλα ζητήματα, παρατηρήσεις Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Συμβιβαστική πρώτη, ένα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 100. 77 υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 187 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3b υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2-2-3, 223 υπέρ κατά αποχές έλεγχος That Απορρίπτεται. Μπορεί μερικές φορές το αποτέλεσμα να είναι με μικρή διαφορά. Θα το ελέγχουμε. 236 υπέρ. Με συγχωρείτε. 235, 235. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Λείπει ένας. Πέρας. Απορρίπτεται. 236. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Κλάς. Πέρας. Απορρίπτεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4α υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Okay, Απορρίπτεται. 12 και 35 που σχεδίονται με τη συμβιβαστική 25. Ε, Οπότε αν καταπέσει θα τις ψηφίσουμε. 47 λοιπόν. M 47 υπέρ. Κατά αποχές. Με συγχωρείτε. M 47 και πάλι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Έλεγχος. Sorry, my mistake. All right. Δικό μου το λάθος. 4-5. 276 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 330 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 29. 364. 364. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 401 τα 401 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Απορρίπτεται. Γιατί είναι ισοψηφία το αποτέλεσμα. 402 και 403. Διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Θα την ψηφίσουμε όταν ψηφίσουμε και την συμβαστική 28. Συμβαστική 9 στη σελίδα 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προστατικό στη συμβαστική 9 υπέρ κατά με συγχωρείτε, να το ξανακάνουμε. Για την προσθήκη, το προσθετικό υπέρ κα... έλεγχος. Είναι ένας υπεράριθμος των σοσιαλιστών. Κάποιος από τους σοσιαλιστές παρακαλώ να μην ψηφίσει. Ίσως κάποιος από τους αναπληρωτές για τους σοσιαλιστές. Είναι ένας παραπάνω. Απορρίπτεται. Όχι, όχι, εγκρίνεται. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε. Ε, ε, το προσθετικό 9 εγκρίθηκε. 444, 444, διαγραφή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η διαγραφή εγκρίθηκε. Παραγραφός 10β, 452, 452 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 453 υπέρ, διαγραφή και πάλι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «464 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 465 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 466 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 467 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 469 υπέρ, 469, 470 και 471 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 488 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθετικός 14α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 395 υπέρ κατά αποχές 496 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 497 υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Και 497 καταπίπτει. 498 498 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Εγκρίνεται. 499. Καταπληκτή. 501. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. απορριπτέ. 500 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω και αυτή απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προστατικό στη συμβαστική 15. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πεντακόσια υπέρ κατά έλεγχος. Από την πρώτη. 546 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ...547 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 548 υπέρ και 549 υπέρ, κατά, έλεγχος. Εγκρίνεται. 550, τροπολογία 550, διαγραφή, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16C, 585, υπέρ, κατά, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. 585 εγκρίνεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 610 υπέρ κατά να ελέγξουμε Αγκρίνεται. 613. Διαγραφή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 18α. Εγκρίθηκε. Προσθετικό προσθήκη στο 18α. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουν τέσσερις επιπλέον. Τέσσερις που δεν θα έπρεπε. Δύο, πέρασαν. Τροπολογία 622. 622 υπέρ, κατά, έλεγχος. Εγκρίθηκε. Όχι, απορρίπτεται. Κουλτ 24. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Εγκρίθηκε. Πουλ 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι μπορείτε τέλος να το ελέγξουμε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18B. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προστατικό 18B. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ο πρόεδρος Μπούζεκ. Ευχαριστώ Βική. Συνεχίζουμε. Τροπολογία υπαριθμών 633. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 634. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 19α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη στην 19α. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 668 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 694 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. The is closed. Rejected. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 697 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 20 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Προστίκη στην 20 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτηκε. Τροπολογία 729 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη στην 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο επαληθεύσουμε. Είναι η πρώτη προσθήκη η πρώτη προστίκη στην Συμβαστική τροπολογία 21. Κλείνει η σοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερη προσθήκη στην 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία. Συμβαστική τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 22. Α νέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 800 υπέρ. Όχι. Τροπολογία 800 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Close. Λήξη της οφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 802 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 803 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπλοκ συμβαστικών τροπολογιών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη 1 στη συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Απο... Ε, επαλήθευση. I close the vote. Λήξη ουσοφορίας. <coughs> Εγκρίνεται. Δεύτερη προσθήκη στην 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. I close. Λήξη ουσοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία, μάλλον προσθήκη στην συμβαστική 25, υπέρ. Κατά. Αποχές, επαλήθευση και πάλι. Addition to compromise 25. I close it. Προσθήκη στην 25. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Amendment. Συμβαστική τροπολογία. Ε, συγγνώμη, τροπολογία 9-19. Υπέρ. 9-19. Υπέρ. Υπέρ. Ετοιμή. Υπέρ λέω. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. I close the vote. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη 1 στην 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, αλλά ας το επαληθεύσουμε καλού κακού. Προσθήκη 1 στη συμβαστική 26. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προσθήκη 2 στη συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Edition 2. Προσθήκη 2 στην 26. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 942 υπέρ. Κατά. Εποχές. Επαλήθευση. 942, I close the vote. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 944 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αλλά ας το επαληθεύσουμε. Επαλήθευση την 944. I close the vote. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 954 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση και πάλι. 954. Λήξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 9.55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 9.55. I close. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 9.69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 969. Καλώς. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 27. Υπέρ. εποχές Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 27α. Υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. Τροπολογία 1034 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1035 υπέρ κατά επαλήθευση 1035 άρχεται η ψηφορία λίγη ψηφοφορία. εγκρίνεται 1040 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 1041. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 1049. I open one. Της 1041. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία παριθμών 28. Έχουμε ε, προφορική τροπολογία. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Ποιο είναι κατά της υποβολής αυτής της ε, προφορικής τροπολογίας. Οι σοσιαλιστές απορρίπτουν όλες τις προφορικές ψηφοφορίε. Οπότε ψηφίζουμε χωρίς την προφορική τροπολογία. Συμβατική πρόταση 28 χωρίς προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1071. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α. Επαληθεύουμε. 1071. vote. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1084 υπέρ. Κατά. Εποχές. Επαλήθευση. 1084. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1157 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 1157. Check. I close the vote. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1185. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1199 υπέρ κατά αποχές ευαλήθευση 1199 I close the door. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 1202. Υπέρ. Κατά. Εποχές Επαλήθευση. close. Λήξη ψηφοφορια Απορρίπτεται 33 α συμβαστική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 33 β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 33 33c υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Προστίκη στην 33 c υπέρ κατά, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προστίκη 2 στην 33 C, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 33 D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1238 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 1242 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 42 Λήξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 35 υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 35α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 36α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1265 υπέρ κατά αποχές ε, παλήθευση 1265 είναι τροπολογία στον κατάλογο ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι λήξη ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1277 υπέρ. Κατά αποχές. Επαλήθευση. 1277. 1277. Απορρίπτεται μάλλον, αλλά το επαληθεύσουμε. να κοιμηθούμε ήσυχα. 1281 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ωραία, επαληθεύουμε. 1281. Λήξη ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 1285 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 0 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. I close Λίγη ψηφοφορία απορρίφθηκε. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση 104 104 λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 146 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. We check electronically. I close the vote. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Εποχές ας επαληθεύσουμε. I close the Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 157. Λήξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 162. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Επαλήθευση. 162. Λήξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 165. Υπέρ. Κατά. εποχές Επαλήθευση. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα, πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 7 και 20. Στις 8 και 20. Στις 8 και 20. Τι, τι λέτε γι' αυτό. Αν ρωτήσετε εμά, μπορούμε να ψηφίσουμε. Βίκυ. Βίκυ είναι υπέρ του να ψηφίσουμε. Ηλεκτρονική, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία, ε, άρχεται. I close the vote. Λήξη ψηφοφορία. 80 υπέρ. Uh, Κυρίε και κύριοι. και κύριοι. Δεν βλέπετε τα χαμόγελα των δύο συγκεκριών μας. Εάν θα έχουν την καλοσύνη να σηκωθούν για να στραφούν προς το ακροατήριο και να τις δείτε. You see, uh, we created in... Βλέπετε ότι καταφέραμε με ένα τεράστιο δυναμικό για συνεργασία και βέβαια έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο νομοθετικό έργο. Έχουμε προετοιμαστεί όμως για εξαιρετική συνεργασία τουλάχιστον μεταξύ έξι κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ θερμά. Ζητώ συγγνώμη αν σας καθυστέρησα και έχετε καμιά συνεδρίαση για τις 8. Μπορείτε να τρέξετε. Αλλά δεν φαντάζομαι να είχατε άλλες δεσμεύσεις. Γιατί έπρεπε να είστε εδώ. Βίκυ Φόρτ. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Καλά Χριστούγεννα και ελπίζουμε τον Ιανουάριο να σα δούμε στην Ολομέλεια με το ίδιο θέμα. Και καλά Χριστούγεννα. Και η συγγήτριά μα θέλει να πει. Οι συγγήτριέ. Αγαπητέ φίλε, θέλετε να πείτε κάτι. Θέλετε να, πει, να μιλήσετε.